Uh, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω την υπογραφή του πακέτου του χρηματοπιστωτικού πακέτου, το οποίο θα αποτελέσει το, υποπτικό το, το εποπτικό μηχανισμό των ε, χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων με βάση την νομοθετική διαδικασία. Υπογράφουμε ένα σύστημα ελέγχου και αξιολόγησης κινδύνου που θα αναλάβει την εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Δεύτερον, δημιουργούμε επίσης τρεις, τρία, τρεις άλλες εποπτικές αρχές για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος που θα παρακολουθούν τις τράπεζες, τη αχρεόγραφα και τις αγορές και τις ασφαλιστικούς οργανισμούς και τις ε, συντάξεις. Και τέλος υπογράψουμε μία οδηγία που συμπεριλαμβάνει 11 οδηγίες με σκοπό να ευθυγραμμιστούν αυτές με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας. Uh, με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας καταβλήθηκαν τεράστιες προσπάθειες με πολύ στενή συνεργασία ε, όλων των ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθήθηκε μια πολύ αποτελεσματική και ταχεία διαδικασία. Οι διαδοχικές προεδρίες, η Ισπανική, η Βελγική, ε, επέδειξαν τεράστιο δυναμισμό. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας και η Επιτροπή δραστηριοποιήθηκε και συνεργάστηκε στενά με τα άλλα θεσμικά όργανα Ευχαριστώ τους, ε, τους συνεργάτες, όλους τους συνεργάτες και όλους τους επιτρόπους που και εκείνοι ανέλαβαν ε, σημαντική δράση σε όλες τις συναντήσεις, σε όλες τις συζητήσεις. Οι συνεργάτες μου, το ίδιο ισχύει και για τους συνεργάτες μου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει τελειώσει η δουλειά μας έχουμε τώρα το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης που το συζητούμε αυτή τη στιγμή που είναι επίσης κάτι το πολύ σημαντικό στα πλαίσια της νομοθετικής μας διαδικασίας και ελπίζουμε ότι θα είναι έτοιμο το ταχύτερο δυνατό. Και ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι αυτά τα έγγραφα που υπογράφουμε σήμερα θα τεθούν σε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου του 2011. Σχεδόν άμεσα δηλαδή. Και αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό για όλους μας και για τις αγορές και για τους πολίτες μας βεβαίως, τους οποίους θέλουμε να βοηθήσουμε. Παρακαλώ λοιπόν όλοι μαζί να υπογράψουμε τα σχετικά έγγραφα.